Καλησπέρα σε όλους, λέει σε διάφορες γλώσσες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Καλησπέρα και σε τελικά, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ερήτημοι συνάδελφοι βουλευτές, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, σας ευχαριστώ που εδώ βρισκόσαστε σήμερα, παρόντες στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που γίνεται επί την ευκαιρία της Παγκοσμίου ημέρας του τουρισμού. Η παρουσία σας και διάφοροι εκπρόσωποι των διεθνών θεσμών, ευρωπαϊκών θεσμών, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης δείχνουν το σημαντικό χαρακτήρα το διατομεακό που έχει ο τουρισμός. Από την αρχή της θητείας μου πρόσπασα να μειώσω την απόσταση που υπήρχε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών, πολλαπλασιάζοντας τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν την συζήτηση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μέσω συναντήσεων για να συζητείτε το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο μέσω μεταξύ των κοινοβουλευτικών, όχι μόνο μεταξύ εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων, αλλά υπάρχει συζήτηση και με τους άμεσους εκπροσώπους των πολιτών, που είναι εκπρόσωποι των ενδιαμέσων φορέων. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ανταλλαγή απόψεων, χρειαζόμαστε μια συζήτηση, άμεση επαφή, συγκεκριμένη για να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες μας. Η δήλωση που στις 25 Μαρτίου στη Ρώμη, στη Σύνοδο Κορυφής, από τους αρχηγούς κρατών κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τα 60 χρόνια της υπογραφής των συνθηκών δείχνει μεταξύ πρώτων προτεραιοτήτων ότι είναι η ανάπτυξη και απασχόληση. Πρώτη στόχη, πρώτη στη. Εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβα την υποχρέωση να εξασφαλίσω το να μην μείνουν άσκηση επιχάρτου αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να πλησιάσουμε του πολίτε. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν συγκεκριμένε απαντήσει ε, σε αυτού και στου διαφόρου φορεί που του εκπροσωπούν. Θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε όλοι να μπορούν να έχουν μια δουλειά, διότι άνευ δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Κανεί δεν θα πρέπει να μείνει πίσω, κυρίω εκείνοι που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τι βιομηχανικέ και τεχνολογικέ επαναστάσει που μεταμορφώνουν τον κόσμο τη παραγωγή και τη παροχή των υπηρεσιών. Αλλάζει η μορφή τη αγορά-εργασία και χρειάζονται οι αναγκαίε δεξιότητε που, αλλάζουν. Δείχνουν μελέτε ότι η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση μπορούν να αντικαταστήσουν σχεδόν το ίμιση τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Μόνο στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύουν περίπου 54 εκατομμύρια θέσει εργασία. Άρα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές για να ρυθμίσουμε τις αλλαγές επενδύοντας περισσότερα και επενδύοντας σε μια κατάρτιση που κρατά το ρυθμό της αγοράς. Όχι μόνο για τους νέους αλλά για όλους τους εργαζομένους που κινδυνεύουν Λοιπόν, παραδείγματο χάρη, όπω αυτοί που ανησυχούσαν, δεν φτιάχνανε τροχού για άμαξε στην παραμονή τη εφεύρεση του αυτοκινήτου. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στην ψηφιακή επανάσταση. Ε, ε, λοιπόν, Λοιπόν, χρειάζεται σύμπραξη με άλλους, με διάφορους τομείς. Ε, βιοτεχνία, ε, γαστρονομία και την ε, χειροτεχνία κλπ. να υπάρχει συνεργασία όλων των τομέων. Θα πρέπει να λάβουμε πλήρως υπόψη το χαρακτήρα, το στατικικό που έχει αυτός ο τομέας. Ήδη σήμερα ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και της απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να καταργήσουμε τις κοινοτοπίες που, που θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικός μόνο για την Νότια Ευρώπη ο τομέας. Και είναι κάτι που ε, και αντιτίθεται κάπως στην ανάπτυξη του τομέα. Λοιπόν, προσελκύεται ο τουρισμός από, ε, από τη βιομηχανία και ανάποδα όχι μόνο για λόγο γαστρονομίας, οπτικοκουστικός τομέας, design, όλα αυτά επηρεάζονται. Λοιπόν, έχουμε προϊόντα αριστείας που παράγονται στην Ευρώπη και κάποιος που βλέπει αυτά τα προϊόντα από το εξωτερικό θέλει να έρθει στις χώρες μας να δούμε. Οι Αμερικανοί ε, που παίρνουν προϊόντα από εμά θέλουν μετά να αγοράσουν τα προϊόντα, έρχονται εδώ, βλέπουν τα προϊόντα και θέλουν να τα αγοράσουν στη χώρα τους. Λοιπόν, έχουμε ένα μοσαϊκό που δημιουργεί επιχειρηματικό ιστό στην Ευρώπη, επικοινόμορφο. Έχουμε διάφορα, διάφοροι τομεί επηρεάζονται, δημιουργική βιομηχανία, κατασκευέ, τουρισμό, ε, ναυπηγεία κλπ. αυτόν τον τουρισμό. Είναι μια βιομηχανία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλου του τομεί, σε όλη την Ήπειρό μα. Λοιπόν, στην Αγγλία και στη Γερμανία ε, έχουμε το 20% από εκείνων που ασχολούνται στον τομέα είναι μικρότεροι από 25 ετών. Λοιπόν, από τα μεγάλα προβλήματα είναι η ανεργία των νέων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτό το στοιχείο ότι απασχολεί πολλού νέου ο τουρισμό. Είναι από τι πρώτε θύρε πρόσβαση στην εργασία ο τουρισμό και είναι συγκεκριμένη ε, απάντηση στην ανεργία. Κυρίω στι νότιε περιοχέ τη Ευρώπη, όπου ένα νέο στου δύο ακόμα δεν βρίσκει δουλειά στην Νότια Ευρώπη. Ε, λοιπόν, σύμφωνα με διάφορου φορού, την επόμενη δεκαετία μπορούμε να δημιουργήσουμε περίπου 5 εκατομμύρια θέσει απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδέονται με τον τουρισμό και το ΑΕΠ θα περάσει από το 1,6 στο 2,13 ευρώ. Αυτό χάρη στην ε, προσπάθεια που θα καταβληθούν μέχρι το 2030. Πάνω από, 2 από 1 στα 2 δισεκατομμύρια θα αυξηθούν οι επισκέπτες από την Ασία. Έχει ιστορική πολιτισμική κληρονομιά και δημιουργική η Ευρώπη και προσελκύει μπορεί να προσελκύσει και να ικανοποιήσει τη νέα ζήτηση. 550 εκατομμύρια αφήξει έχουμε σήμερα και είμαστε ο πρώτος προορισμός των τουριστών. Το 2020 μπορούμε να πετύχουμε τα 700 εκατομμύρια, φτάσουμε τα 700 εκατομμύρια. Θα ήταν σοβαρό σφάλμα αν οι πολιτικοί θεωρήσουν ότι εκ Θεού ε, θα δημιουργηθεί αυτή η αύξηση. Χρειάζεται προσπάθεια. Συναθηνά Αθηνά και χειρακίνη. Λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο. Λοιπόν, δείχνουν οι προβολές το 2030 λιγότερο το 1 τρίτο των τουριστών ε, θα έρθει στην Ένωση. Αυξάνεται η παγκόσμια, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, ε, υπάρχουν ανταγωνιστικές τιμές, νέοι προορισμοί. Πρέπει να κινηθούμε. Για να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη δυνατότητα τομέα θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί βασιζόμενοι στην ποιότητα και την βιωσιμότητα. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να επεξεργαστούμε τέσσερι πυλώνε. Πρώτον, να προσελκύσουμε περισσότερε επενδύσει, αυξάνοντα και κάνοντα πιο αποτελεσματική την χρήση των πόρων των κοινοτικών και βελτιώνοντα ε, το όλο πλαίσιο τη επιχειρήση. Δεύτερον, να έχουμε προωθήσει μια κατάρτιση που αντιστοιχεί στι ανάγκε του τομέα. Ε, τρίτον, χρειάζεται καλύτερη διακυβέρνηση και χειρισμό τη ψηφιακή επανάσταση. Τέταρτον, να εκμεταλλευτούμε διάφορε συμπράξει για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να προωθήσουμε την Ευρώπη στι ε, διεθνεί αγορέ. Ξεκινώντα βέβαια από την Κίνα. Ο τουρισμό ε, πρέπει να περάσει διάφορα εμπόδια. Θα τα αναφέρουν άλλοι. Έχουμε υψηλή φορολόγηση σε χώρε, άμεσου φόρου, έμεσου φόρου που στην Ευρώπη βαρύνουν περισσότερο από αλλού τον τομέα. Κόστος μεταφορικό, ενέργεια, η έλλειψη των υποδομών είναι προβλήματα, όπως ευρυζωνική ε, παροχή ε, υπηρεσιών στην Ήπεθρο κλπ. Και τοπική, ε, τοπικές μεταφορές. Η πρόσβαση στις πιστώσεις είναι ένα άλλο πρόβλημα. Οι πολιτικοί σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να λύσουν αυτούς τους γόδιους δεσμούς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε βιώσιμο τουρισμό μέσω επενδύσεων για να αυξήσουμε ε, ενεργειακή απόδοση, και καινοτόμε πηγέ ενέργεια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στατικέ Επενδύσει. Αυτέ οι επενδύσει πρέπει να γίνουν, θα αποπληρωθούν σε κάποια χρόνια και θα γίνει ο τουρισμό ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστικό και θα βοηθήσει στο ε, να, να πετύχουμε και του στόχου που έχουμε για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Δεν πρέπει να περιοριστούμε όμω τη βιωσιμότητα του τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να προσελκύσουμε και πόρου για να βελτιώσουμε τη διασυνδεσιμότητα, τη ψηφιοποίηση των μουσείων, τη διασυνδεσιμότητα των αερο, ε, αεροδρομίων κλπ. Καλύτερη χρήση των περιφερειακών πόρων πρέπει να γίνει και του ορίζοντα 2020 σε συνεργασία με τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τις επενδύσεις. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη διάδοση να χρησιμοποιήσουμε τη διάστατη απεικόνηση ε, στα διάφορα μουσεία, ε, να προβάλλουμε του αρχαιολογικού θησαυρού και την ιστορία μα χρησιμοποιώντα την τεχνολογία με τη διάστατη προβολή κλπ. Ε, μπορούμε βάσει προγραμμάτων πιλωτικών να προσελκύσουμε, όπω στην Ακρόπολη, να προσελκύσουμε όπω είναι η Πομπία, η Κνωσό, το Κολοσσέο, όλα αυτά να προβάλλονται τρισδιάστατα. Όπω παλαιολιθικέ πηγέ στην Ισπανία και στη Γαλλία, για να προσελκύουμε τουρίστε. Ο νέο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, πρέπει να λάβει υπόψη τι ανάγκε των πολιτών περισσότερο, όπω είναι η καταπολέμηση τη ανεργία. Λοιπόν, θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο την προσέλκυση επενδύσει για έρευνα και καινοτομία. Θα πρέπει να σκεφτούμε και μια ιδιαίτερη πρικοδότηση για τον τουρισμό, κάτι που ζητήθηκε το 2015 από την έκθεση De Monti, που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη κάναμε κάποια πράγματα με το πακέτο κόσμου αλλά έχουμε ε, αιτήσει που απορρέουν από την έκθεση Τεμόντι που είναι ακόμα πιο φιλόδοξε απαιτήσει. Ε, χρειάζεται να απελευθέρωσουμε και του επιχειρηματίε από τη γραφειοκρατία που πολύ συχνά είναι άχρηστη και επαχθής αυτή η γραφειοκρατία. Η οδηγία των υπηρεσιών δεν έχουμε στόχο να διευκολύνει μόνο ψηφιακέ πλατφόρμες αλλά να βελτιώσει την αδειοδότηση για τι επιχειρήσει. να τις κάνει πιο ανταγωνιστικέ. Επαγγελματική κατάρτιση. Άλλο ένα στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να έχουμε νέους που θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα σημερινά. Είπαμε πώς θα πρέπει να βελτιωθεί ο τομέας της βιομηχανίας του τουρισμού και αν εμείς δεν βασιστούμε επί των νέων, επί της κατάρτισης των νέων, δύσκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα ε, μία από τη σχολή που προάγει την αριστεία, τη Φεράντη για την αστρονομία. Και εκεί ε, ε, εκπαιδεύονται νέοι που είναι έτοιμοι να κινηθούν στον τομέα του τουρισμού σε κάθε επίπεδο. Από τον απλούστερο τομέα μέχρι τον πιο περίπλοκο. Ευχαριστώ και τους Επιτρόπους Μπιενκόφσκα και, και Τίσεν που εισήγαγαν τον τουρισμό, Μπιενκόφσκα μάλλον, συγγνώμη, στα πλαίσια του θεματολογίου για τις δεξιότητες μέσω συγκεκριμένων ειδικών πόρων για αυτόν τον σκοπό. Θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ο επόμενο προπολογισμό θα πρέπει να ε, θαρρύνει την κατάρτιση, ούτω ώστε η μαθητεία να μπορεί να φτάνει και μέχρι τα 25 έτη. Θα πρέπει ε, να υπάρχουν ε, μέσω του Εράσμου διασυνοριακέ προσπάθειε και το Έρασμο για του νέου επιχειρηματίε πρέπει να προωθηθεί. Λοιπόν, μετά Μπορεί αυτοί που πηγαίνουν το χειμώνα στις Άλπες, στις Άλπες, ε, στη Γαλλία και την ε, Ιταλία μπορούν μετά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Ισπανία και την Ελλάδα το καλοκαίρι. Μετά έχουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες, ένα άλλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να υπάρχουν κανόνες ε, διαφορετικοί από, για εκείνους που κινούνται εντός και εκτός του, του διαδικτύου. Οι πλατφόρμες έχουν γίνει νόμος έχουν δεσπόζουσα θέση επί της αγοράς και δίνουν ελάχιστους φόρους και μεταθέτουν μεγάλο πλούτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες του κόσμου αυτές οι πλατφόρμες, όπως η Google. Δεν έχει τις υποχρεώσεις για την προστασία του copyright και των ανηλίκων, ε, ενώ ε, μαζεύει πολλά λεφτά από τις ε, πολλές διαφημίσεις. Και τι συμβαίνει, αυτές οι διαφημίσεις που προέρχονται και από γίγαντες που ελέγχουν το 90% των κρατήσεων online και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων, ε, μειώνοντας το περιθώριο κέρδος αυτών, ε, αυτοί ε, βγάζουν τα κέρδη άλλα, και δρεύουν σε άλλα μέρη του κοσμού και δεν δημιουργούν ούτε πλούτο ούτε απασχόληση στην Ευρώπη. Τα ίδια ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τι πλατφόρμες αυτές. Και δεν πληρώνουν αρκετού φόρου οι πλατφόρμες. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Πρέπει στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων να καταλήξουμε σε φορολογική εναρμόνιση που θα επιτρέψει να προσπιστούμε και την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης, που είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, ουσιώδες, ε, της πολιτικής που ακολουθούμε για τον τουρισμό. Η καλά έκανε Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επέβαλε κυρώσεις στην Google, διότι δεν σεβάστηκε η Google τους κανόνες που οι άλλοι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σέβονται. Και η συνεργατική οικονομία. Έχουμε δύο τέτοια πρότυπα αυτού του νέου μοντέλου επιχειρήσεως. Ε, το Uber και τα Bread and Breakfast ε, που βλέπουμε που έχουν προωθηθεί. Οι ανταγωνιστέ του στη μεταφορά, την τοπική μεταφορά, πρέπει να σέβονται όμω προδιαγραφέ στου εργαζομένου, του καταναλωτέ για την ασφάλεια κλπ και συνθήκες αδειοδότησης που επηρεάζουν πολύ λίγο όμως τους γίγαντες του τομέα. Θα πρέπει και τους δίνουν πλεονέκτημα. Ξέρω ότι οι, επίτροπος, οι διάφοροι ομάδες επίτροποι επεξεργάζονται το θέμα αυτό για να δημιουργήσουν πραγματική ε, αγορά για υπηρεσίες και ψηφιακό τομέα. Η αγορά της Ένωσης πέρα που πρέπει να προωθηθεί την καινοτομία και την οικονομία κλίμακα, πρέπει να έχει κανόνε ανταγωνισμού και πρέπει να επικρατεί ισοτιμία όσον αφορά τι συνθήκε που ισχύουν για όλου. Θα πρέπει, λέγω κλείνοντα, να προωθήσουμε μαζί την Ευρώπη σαν πρώτη στο προορισμό τουριστικού στον κόσμο. Το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς και, αυτός και το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, Κίνας. Τον επόμενο χρόνο, 19 Ιανουαρίου, έχουμε τέτοια σύνοδο κορυφή σε ένα φόρουμ στην Βενετία για την προώθηση του θέματο συμμετοχή επαγγελματιών τη Βενετία ε, και τη Κίνα, τη Ευρώπη και τη Κίνα. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο τη Βενετία και τον Επίτροπο Μπιενκόφσκα και τον Επίτροπο Ναύρα Σίτ για τι προσπάθειε που καταβάλουν για την υλοποίηση αυτή τη ε, πρωτοβουλία. Ιδιαίτερα χαίρομαι σήμερα και για την παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO Ερίνα Μπουκόβα, της κυρίας Μπουκόβα. Στη 18 θα έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε, το 18 θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την πολιτισμική μας διπλωματία έχοντας πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν εκεί για ανάπτυξη και απασχόληση που απορρέουν από την εκμετάλλευση του πολιτισμικού μας τομέα και της δημιουργικότητας. Πρέπει να έχουμε περισσότερους διεθνείς τουρίστες που θα πρέπει να προωθούμε συνολικά την Ευρώπη σαν έναν προορισμό όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και τον Καναδά. Ένας Κινέζος επισκέφτεται 4-5 κατά μέσο όρο. Ο ανταγωνισμός δεν είναι μεταξύ Γαλλίας, Ισπανίας ή περιοχών της Ιταλίας. Επιλέγει πάνω από όλα την Ήπειρο ταξιδιώτης που θα πάει. Όπου πρέπει να, να πάμε εναντίον Αμερικής, Ασίας, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές μας. Όποιο αποφασίζει να πάει να κάνει σκι στι Άλπε ή να κάνει κουαζιέρα στη Μεσόγειο, επιλέγει την Ευρώπη. Και εμεί θα πρέπει να δώσουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κλειδιά, αν θέλετε, για να ανοίξουν οι πόρτε. Και μετά να αρχίζουν να τριγυρνάνε αυτοί οι άνθρωποι εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μπορεί να μπει κανεί στη Γαλλία, γιατί τον προσελκύει η γαλλική γαστρονομία. Μετά να πάει προς τη Γερμανία, μετά μπορεί να πάει από τη Γερμανία στην Ουγγαρία, μετά από την άλλη πλευρά της Ευρώπης να πάει να Ισπανία, Ισπανία Πορτογαλία. Όποιος ε, συνηθίζει να ταξιδεύει 15-20 μέρες μπορεί να κάνει αυτού του είδους τα ταξίδια και το πρώτο κλειδί βοηθά να ανοίξουν και άλλες πόρτες. Πιστεύω ότι στον επόμενο προϋπολογισμό χρειάζεται ένα ταμείο, ένα πόρο τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να ενεργοποιήσουμε συγχρηματοδότηση τουλάχιστον ε, για, από πλευρά τοπικών αυτοδιοίκησεων. Αυτοί οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πολλαπλασιαστούν με τη συνεισφορά των διαφόρων και θα προσελκύσουμε από τον υπόλοιπο κόσμο τουρίστε και να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Έχουμε ήδη μια σειρά τουριστικών προϊόντων ε, και τραστ που έχουμε προωθήσει από Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τα, τα δίκτυα της UNESCO και λοιπά και τα πολιτισμικά, τις πολιτισμικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης ή το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό που στηρίζεται από τον Επίτροπο Μπέλα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους βουλευτές, τους συναδέλφους, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα ήταν ενεργό να κινητοποιεί να παρακινεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιεί πιο ε, ενεργέ πολιτικές στον τουρισμό. Και αυτό σε χάρη σε κάποιου βολητέ που θα ε, που ε, συμμετέχουν στην Task Force και στην ομάδα, κομματική ομάδα για τον τουρισμό και στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών. Υπάρχουν και κάποια προγράμματα το, Ευρωπαϊκή, το έντος Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κίνας, διάφορες φωτοβουλίες, τα πολιτιστικά μονοπάτια, διαδρομές και το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του, ε, ε, του τουρισμού που από το 2020 θα ξεκινήσει. Λοιπόν, στις 29 Οκτωβρίου του 2015 είχαμε υιοθετήσει ένα ψήφισμα πρωτοβουλίας όσον αφορά τις νέες προκλήσεις για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Το έγγραφο υπογραμμίζει την ανανεωμένη ε, σημασία που έχει ο τουρισμός που αναφέρεται συνθήκη της Λισαβόνας και ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε κατάλληλη στατική για την Ευρώπη. Ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ο πρώτος προορισμός στον κόσμο. Ε, να δώσουμε νέα όθηση στον τουρισμό τον ευρωπαϊκό. Το 2010 ξεκινήσαμε όλα αυτά. Λοιπόν, ε, είναι σαφή η θέση του Κοινοβουλίου. Ο τουρισμό δημιουργεί ανάπτυξη, απασχόληση, επενδύσει και ανάπτυξη των περιοχών. Γι' αυτό τα θεσμικά όργανα τη Ενώση πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερο, ώστε να προωθήσουν μια προσέγγιση συντονισμένη μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κρατών Μελών και τοπική αυτοδιοίκηση και βιομηχανία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στρατηγική που θα ενσωματώνει το, τον τουρισμό και θα το συμπεριλαμβάνει στον επόμενο προπολογισμό. Να αξιολογήσει επίση και το αντίκτυπο που έχουν άλλε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω επί του τουρισμού, ξεκινώντα ε, από την ολοκλήρωση τη αγορά των υπηρεσιών και τη ψηφιακή αγορά. Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε την Παγκόσμια Μέρα του Τουρισμού για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση όσον αφορά τον αυτού του τομέα. Σήμερα είναι η μέρα φιλοδοξίας, θάρρου νέων προτάσεων που θα πρέπει να έχουν στόχο να ξεπεραστούν σημαντικά όρια. Αν συνεργαστούμε όλοι, ο διπλασιασμό των αφήξεων την επόμενη δεκαετία δεν θα είναι απλώ ένα όραμα, μια αυταπάτη. Και σκεφτείτε πώ θέσει εργασία μπορούν να δημιουργηθούν με ένα δισεκατομμύριο ταξιδιώτε εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά χρειάζεται μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική που δεν θα πρέπει να αντιτίθεται με τι στρατηγικέ τι περιφερειακέ ή εθνικέ. Θα πρέπει να ενισχυθούν ή εν λόγω προσπάθειες. Χρειάζεται πραγματικά μια στρατηγική που παρουσιάζει την Ευρώπη σαν ένα κόσμημα που δεν μπορείς να αρνηθείς να το επισκεφθείς, διότι εντός αυτού του κοσμήματος υπάρχουν πάμπολα στοιχεία φωτεινά που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να μη σκεφτεί ότι δεν θα πάει να τα ανακαλύψει. Ευχαριστώ πολύ και καλές εργασίες σας εύχομαι. Καλή δουλειά. Δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριο Κατάινεν. Ε, πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι υπουργοί, πάντοτε αποτελεί χαρά μου να ε, συμμετέχω εδώ στις εργασίες του Κοινοβουλίου και ειδικότερα με αυτόν τον πρόεδρο ο οποίος βέβαια ήταν αρμόδιος ε, στο παρελθόν από πλευρά και της ε, Επιτροπή ε, για τα ζητήματα και του τουρισμού και τη απασχόληση. Και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού. Πρόκειται για έναν τομέα όπου έρχονται από τον οποίο προέρχονται διάφορες καινοτομίες. Και ο τουρισμός έχει ε, μία σειρά από πλεονεκτήματα, soft όπως τα λέμε, δηλαδή όχι ιδιαίτερα Ε, δηλαδή, ε, η, τα έθι, η ήθη και τα έθιμα είναι εκείνα τα οποία αξιοποιεί ο τουρισμό και τα οποία έχουν οικοδομήσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επίση, ο τουρισμό είναι ένα κλάδο ο οποίο συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αποτελεί δηλαδή την ε, οικονομική κινητήρια δύναμη για μία σειρά από περιοχέ τη Ευρώπη. Ε, πέρυσι, ε, συνεισέφερε ο τουριστικός κλάδος ε, κατά 10% ε, στο συνολικό ΑΕΠ ε, της Ένωσης με ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 3%. Οι επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, στον τουρισμό δημιουργούν, ανάπτυξη δημιουργούν θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις αποτέλεσαν την καρδιά του θεματολογίου της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή η προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης αποτελούν κύριες προτεραιότητες από τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής. Και γι' αυτό πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε ε, αυτό το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής σε αυτό το ε, σχέδιο. Ε, ο στόχος μας ήταν να αποδεσμευτούν 350 δις επενδύσεων στον τουριστικό τομέα έως το 2018 και ήδη μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε 236 δισεκατομμύρια επενδύσεις σε αξία, ειδικότερα σε μικρής ε, κλίμακας ε, ε, project, έργα δηλαδή, σε μία σειρά από διαφορετικά κράτη-μέλη. Και ε, ε, στην κοινή ε, συνεδρίαση που έγινε μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπή αποφασίστηκε να πρικοδοτηθεί περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τι Στρατηγικέ Επενδύσει, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί με αυτέ τι σημαντικέ συμπληρωματικέ επενδύσει θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερη ανάπτυξη, ακόμα περισσότερε εργασίε και περισσότερη ανταγωνιστικότητα συμπεριλαμβανομένου και του τουριστικού κλάδου. Και στον σχετικό κανονισμό αναφέρεται και ρητά ο τουρισμός ε, ω ένας από τους τομείς ο οποίο μπορεί να λάβει τέτοια έργα από το ΕΦΣΕ. Και εδώ βέβαια αναφερόμαστε σε έργα τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα σε όλες τις περιοχέ τη Ένωση. και υπάρχουν μια σειρά από δυνατότητες. Ε, για παράδειγμα, οι δράσεις, ε, οι επιλέξιμες στον τομέα του τουρισμού αφορούν για παράδειγμα την ενεργειακή αποδοτικότητα ξενοδοχείων, είναι την ζωγόνηση κάποιων εκτάσεων για τουριστικούς σκοπούς ή και χρηματοδοτήσεις, συμφωνίες χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, τα έργα τα οποία μπορούν λοιπόν να επιλεγούν για χρηματοδότηση μπορούν να λάβουν χώρα σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να έχουν και διασυνοριακό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κάποια ποσόστοση γεωγραφική σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους έργα που μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Και για να σα δώσω ένα παράδειγμα ω προ το τι μπορεί να υποστηρίξει και πώ μπορεί να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο, το ΕΦΣΙ, θα σα δώσω κάποια παραδείγματα. Στην Ελλάδα το ΕΦΣΙ ήδη υποστηρίζει ε, την αναβάθμιση τριών περιφερειακών αεροδρομίων. Πράγμα βέβαια το οποίο θα αναβαθμίσει το προφίλ της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό και αυτό με τη σειρά του θα συμβάλλει στο αναπτυξιακό δυναμικό στο σύνολο της χώρας. Στην Πολωνία το ΕΦΣΙ ενισχύει μια επιχείρηση η οποία ε, δραστηριοποιείται στο ποταμό βίστρο ούτω ώστε να συμβάλλει με τη σειρά τη στην ε, ανάπτυξη. Πράγμα το οποίο βέβαια ήδη οδηγεί σε αύξηση ε, της οικονομικής δραστηριότητας τη επιχείρηση αυτή κατά 15-20%. Στη Σουηδία είχαμε μία χρηματοδότηση η οποία αφορά αποκλειστικά στην κράτηση online για άτομα τα οποία έχουν ε, κάποια ε, αναπηρία. Και ε, ήδη ανακοινώθηκαν ότι θα υπάρξουν μία σειρά από περαιτέρω τεχνικέ βελτιώσει σε αυτό το σύστημα κρατήσεων, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν δυνατά μέσω του ΕΦΣ. Επίση, θα ήθελα να τονίσω την σημασία των περιφερειών σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο τη Επιτροπή και θα σα αναφέρω ε, δύο από τα project τα οποία λαμβάνουν χώρα ε, στα ε, υπερπόντα εδάφη της Γαλλίας. Έχουμε λοιπόν εδώ σε τουριστικά project αλλά και επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχουμε μία σειρά από πολύ χρήσιμα έργα στον τουριστικό τομέα τα οποία ήδη έχουν λάβει υποστήριξη από το επενδυτικό μας σχέδιο. Ωστόσο, πάντοτε θα πρέπει και πάντοτε είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό που έχετε ε, κατά νου είναι η δημιουργία πλατφορμών στον τουριστικό κλάδο. Για παράδειγμα, αυτές οι πλατφόρμες θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν ε, τέτοια project αναζωογόνησης, πράγμα το οποίο θα ε, ήταν προς όφελος ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ε, πρόσφατα δημοσιεύσαμε έναν οδηγό πέντε βημάτων σε ό,τι αφορά τη δημιουργία τέτοιου είδους πλατφορμών. Οπότε ελπίζω όλοι σας, είτε εκπροσωπείτε κάποιο περιφερειακό φορέα, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό φορέα, θα ρίξετε μια ματιά σε αυτόν τον οδηγό ω προς το πώ μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια επενδυτική πλατφόρμα ώστε να συνενωθούν τροποντινά μία σειρά από διαφορετικά μικρής κλίμακας ε, project. Κάτι ακόμα που προσπαθούμε εδώ να εξετάσουμε είναι το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την υποστήριξη του ΕΦΣΥ ε, με την χρηματοδότηση από άλλα ταμεία μεταξύ αυτών και τα διαρθωτικά. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ε, υλοποιηθούν project τα οποία δεν θα μπορούσαν σε διαφορετικό τρόπο να υλοποιηθούν. Και η Επιτροπή συνεχίζει να προωθεί και έχει προτάσεις για αυτό το συνδυασμό ΕΦΣΙ και άλλων ταμείων. Τώρα, ο δεύτερος πυλώνας του επενδυτικού ε, σχεδίου αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία, τα οποία ήδη αποφέρουν αποτελέσματα. Το πρώτο από αυτά είναι ε, το ΧΑΠ, το κέντρο, δηλαδή ο κόμβος ε, για τις επενδύσεις και τις πληροφορίες, που παρέχει υποστήριξη στους δημόσιους εφόρες. Και αυτό το αυτός ο κόμπος για ε, τις συμβουλές και τις επενδύσεις ήδη λειτουργεί πολύ καλά με 500 αιτήματα που ήδη έχει λάβει για ε, ε, για παράδειγμα τεχνική αρρωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα των έργων που εκτελούνται ή για παροχή πληροφοριών σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό της χρηματοδότησης από διαφορετικά υφιστάμενα ταμεία της Ένωσης. Και το σημαντικό είναι εδώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει κάποια συμβουλή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ε, περάσουμε στους δυνητικούς επενδυτές αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ε, επιθυμούν να λάβουν βοήθεια. Το δεύτερο τώρα στοιχείο του δεύτερου ε, πυλώνα είναι το project portal όπως λέγεται για τις επενδύσεις. Εδώ μιλάμε για έναν χώρο που συναντούνται οι ενδιαφερόμενοι και οι δυνητικοί επενδυτές. Και εδώ βλέπουμε μία σειρά από project τα οποία εδώ επιδεικνύονται από μία σειρά από χώρες Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Γαλλία, Οπότε θα σας καλούσα όλους να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το πόρταλ και ειδικότερα να το αξιοποιήσετε. Κυρίες και κύριοι, ο τουριστικός κλάδος έχει πραγματικά ένα φανταστικό ε, δυναμικό σε ό,τι αφορά την καινοτομία και παρέχει σταθερή οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Και όχι μόνο μας δημιουργεί τέτοιου τους οικονομικά ε, πλεονεκτήματα, αλλά μας επιτρέπει να φέρουμε πιο κοντά μεταξύ μας τις πολιτισμικές μας ε, ε, κληρονομιές στο πλαίσιο της διαφορετικότητας μας. Και αυτή η ισχύση του τουρισμού είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε ποτέ. Και θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παίκτη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου τη Ευρώπη. Η δική σα δηλαδή στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική για να συνεχίσει να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτέ τι προκλήσει και να παραμείνει ανταγωνιστικό ο ευρωπαϊκό τουρισμό. Α συνεχίσουμε λοιπόν ε, την άγουσα την οποία ήδη έχουμε ε, ξεκινήσει και α συνεχίσουμε περισσότερε επενδύσει μέχρι την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη στράτευσή σας στο πλευρό του τουρισμού που είναι τόσο κρίσιμος για την ανάπτυξή μας. Επόμενη ομιλήτρια είναι επίτροπος ε, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. κυρία Πιανκόσκα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, επίτροποι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι των διαφόρων κρατών μελών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα από την Πολωνία. Σας χαιρετώ. Ε, Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, διάσκεψη αυτή υψηλού επίπεδου για να γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ανέλαβα να σας διαδεχτώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, μου ζητήθηκε υπό την ιδιότητα αυτή να σας πω ότι κάνουμε. Βεβαίως είναι πολλές οι προκλήσεις και στον κλάδο αυτό, αλλά όπως γνωρίζετε μόνο ένα προτεραιότητα της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο και το σωστό κλίμα για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Και πιστεύω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι πολύ σημαντικό και για κλάδους όπως είναι ο τουριστικός διότι ο τουρισμός έχει περάσει ε, τα ίδια δεινά ε, και πλήγματα με την υπόλοιπη οικονομία, αλλά έχει πληγεί διπλά και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την πολιτική αστάθεια γενικώ. Ποια είναι όμως τα καλά νέα και το είδαμε από την ομιλία του κυρίου Κατάινεν. Ε, ανθίσταται ο, ο τουρισμός ε, στην Ευρώπη και αναπτύσσεται και αλλάζει ετώνησε ε, ο Γύρκη ε, πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του τουρισμού στην Ευρώπη στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Περίπου 500 εκατομμύρια ξένους τουρίστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ηγέτης, είναι ο υπαριθμόν ένα τουριστικός προορισμός. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τις πολλές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει και ο κλάδος αυτός. Η σημερινή διάσκεψη εστιάζει στα σημαντικότερα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι επενδύσεις παραμένουν πολύ χαμηλές και αυτό το συνδέω με την ομιλία του Γύρικη Κατάινεν. Δεύτερον, ο τουρισμός ε, χρειάζεται επαγγελματίες με πάρα πολύ καλά προσόντα, ε, διαφορετικά ψηφιακά, διαπροσωπικά, γλωσσικά, επιχειρηματικά, διευθυντικά. Επίσης υπάρχει ψηφιακή και τεχνολογική επανάσταση που ε, καθορίζει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο τουρισμός και δίνει και νέες ε, δυνατότητες για τους ε, πελάτες μας. Έχουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, συνεργατική οικονομία, η οικονομία του διαμοιρασμού. Να σας αναφέρω μερικά στοιχεία και μόνο η Ευρώπη ανταγωνίζεται για να έχει μερίδιο αγοράς με αναδυόμενες ε, αγορές, ιδιαίτερα από την Ασία και τον Ειρηνικό. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε με περιορισμένε νομικέ αρμοδιότητε στον τουρισμό, αλλά θέλουμε πραγματικά να υποστηρίξουμε τον κλάδο, ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις προκλήσεις. Πρώτα, για τι επενδύσει, εργαζόμαστε έτσι ώστε ε, να έχουμε πιο ισχυρές ΣΔΙΤ, ε, συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα και πιο ευφύ χρήση των κοινοτικών πόρων, μέσων και κονδυλίων. Θέλουμε όσο μπορούμε να επενδύσουμε και να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Θα ήθελα να πω και με την προηγούμενη εμπειρία μου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαπεριφερειακή συνεργασία. Έχουμε πλατφόρμες για την ευφύ e, εξειδίκευση, για τον εξυγχρονισμό της βιομηχανίας και ε, σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ελπίζω αυτό το εργαλείο για να διευκολύνουμε τη συνεργασία του κλάδου του τουρισμού με τις περιφέρειες και την ΣΟΤΑ. Επίσης, ενθαρρύνουμε επενδυτικά προγράμματα με μεικτή χρηματοδότηση, κοινοτική, ενωσιακή και ιδιωτική. 70 περιφέρειες έχουν ε, μπει στο πρόγραμμα με 11 θεματικές ε, πλατφόρμες και δίκτυα και με χαρά ε, σας ανακοινώνω ότι μόλις σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε το πρώτο δίκτυο και ανακοινώθηκε. Και το πρόγραμμα COSME ε, μας βοηθάει να υποστηρίξουμε πιο μικρά διασυνοριακά ε, έργα. Για τα προσόντα και τις δεξιότητες. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο. Έχουμε το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες, ε, για τη συνεργασία και πλατφόρμες για τις συγκεκριμένες μορφές τουρισμού είναι ένα προσχέδιο συνεργασίας τομεακής για να δούμε ποια προσόντα και ποιες δεξιότητες χρειάζεται η βιομηχανία. Πολλοί είναι οι τομείς, 7 είναι στην αρχική φάση, αλλά ο τουρισμός επελέγει ως ένας από τους 7 για να δούμε τι χρειάζεται ο κλάδος για να παραμείνει ανταγωνιστικός. Ένα τρίτο σημείο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις να ακολουθούν τις τεχνολογικές και ψηφιακές ε, αλλαγές. Με τη στρατηγική για την ψηφιακή αγορά έχουμε ειδικά ε, σεμινάρια εκδηλώσεις, σεμινάρια στο διαδίκτυο ε, και την πύλη, τη δικτυακή για πώς εφαρμόζεται στον κλάδο αυτό ο Ευρωπαϊκός Νόμος. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν ε, ανταλλαγή καλών και βελτίστων πρακτικών και εμπειριών. Και εσείς του τουριστικού κλάδου ζητήσατε ιδιαίτερη βοήθεια κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του τουρισμού και προτίθεμαι να διοργανώσω διάφορα σεμινάρια, εργαστήρια ακριβώς για αυτά τα ε, θέματα του τουρισμού με τα κράτη-μέλη. Τώρα, ποια είναι η βασική μου ε, ιδέα και πώς αντιλαμβάνομαι το εγχείρημα αυτό να μην εθελοτυφλούμε απέναντι σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό να γίνεται με τρόπο υπεύθυνο, βιώσιμο, με πλήρη σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια συνεργαζόμαστε με τον κλάδο και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής και γενικά για να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε ε, την Ευρώπη σε τρίτες χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Ταξιδίων για να προάγουμε και να προβάλλουμε ε, την κληρονομιά μας, την πολιτισμική, την αρχαιολογική, την τουρισμική του χρόνου. Ε, θα έχουμε το έτος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και θέλουμε να ενταθούν οι τουριστικές επαφές και οι επισκέψεις. Και ε, χαίρομαι που έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων υψηλού επίπεδου με πρώτη αυτή που θα δεξαχθεί στις 19 Ιανουαρίου στη Βενετία. Και πάλι λοιπόν Θέλω να τονίσω ότι έχουμε περιορισμένες νομικές δυνατότητες, αρμοδιότητες όσο και ρόλο, αλλά το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό εργάζομαι με τόσο πάθος, ε, είναι συνεργασία. Διοργανώσει σαν τη σημερινή είναι πολύτιμε. Διάφορα θεσμικά όργανα, δημόσια όργανα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται με τον κλάδο, τα κράτη-μέλη τη περιφέρεια, του δήμους και τι κοινότητε και οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι και παραμένει ένα βασικό ε, πρωταγωνιστής, γιατί η πολιτική σας υποστήριξη και η δική σας προσωπικά πρόεδρε είναι πολύτιμη για μας. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξη πραγματικά για το μέλλον του τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη. Είμαι βέβαιη ότι η τουριστική βιομηχανία μπορεί να είναι και νικηφόρα και ε, ηγέτης στην οικονομία, αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ελπίζω να είστε κοντά μας και στις 28 Νοεμβρίου, που είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού σας εύχομαι καλή συνέχεια και πολύ ε, γόνιμες εργασίες στη διάσκεψη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, κυρία Βιανκόφσκα. Η Γενική Διευθύντρια UNESCO, η κυρία Μπόκοβα. Είχατε το λόγο, κυρία Μπόκοβα. Αξιότιμε ε, κύριε Ταγιάννη, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμε Υπουργοί, Επίτροποι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Σιτήρη. Με τιμή μου, ε, έρχομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ε, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στον τουρισμό της Ευρώπης. Η νέα στρατηγική για τον τουρισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αξία του τουρισμού ω κινητήρια δύναμη τόσο για τη δημιουργία θέσεων εργασία όσο και για την βιωσιμότητα για την οικονομική ανάπτυξη και την ε, κοινωνική ένταξη, την ευρωπαϊκή αυτοεκτίμηση και την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και αυτή η στρατηγική έρχεται σε ένα κομβικό σημείο ε, και έχει σχετίζεται πάρα πολύ με, τις, με τη δική μας εντολή. Σήμερα 1,2 δισεκατομμύρια άτομα διέρχονται διεθνή σύνορα κάθε χρόνο και αναμένεται πως θα αυξηθούν στα 2 δισεκατομμύρια έως το 2030 με τα μνημεία λοιπόν παγκόσμιας μας πολιτιστικής κληρονομιάς, τις ε, προστατευόμενες περιοχές βιόσφαιρας και τα γεωπάρκα της, ε, που αποτελούν και πολλά από αυτά τουριστικούς προορισμού, η UNESCO παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ε, επανάσταση στον τουρισμό. Ο πολιτιστικό τουρισμός αντιποκρίνεται σήμερα στο 40% του παγκόσμιου τουρισμού και με περισσότερα από 300 μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ πλούσια σε, σε αυτήν την κληρονομιά και ε, προφανώ θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την αυξανόμενη ζήτηση από πολλέ σημαντικέ αγορέ, ειδικότερα την ε, Κίνα. Και ο βιώσιμο ε, τουρισμό μπορεί να μετασχηματίσει αυτήν την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά σε μια μοναδική πηγή καινοτομία, δημιουργικότητα και ανάπτυξη. Ε, γνωρίζουμε όμω και πάρα πολύ καλά του ε, κινδύνου τη κακή διαχείριση, κακοδιαχείριση του, τουρισμού και τον αντίκτυπο δηλαδή που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Και φέτο ε, γιορτάζουμε το Διεθνέ Έτο για ε, τον ε, βιώσιμο τουρισμού για την ανάπτυξη και ε, το επόμενο έτος θα εορτάσουμε το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Κίνας όπως και το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. και θεωρώ πάρα πολύ ε, θετική αυτή την ε, απόφαση από την πλευρά, την πρόταση μάλλον του Κοινοβουλίου που έγινε δεκτή. Ε, γιατί θεωρώ πως πραγματικά με αυτόν τον τρόπο ο τουρισμός έρχεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού οράματος τόσο το 2018 όσο και μετά από αυτό. Και πραγματικά θεωρώ πως η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν φυσικούς εταίρους σε αυτό το τομέα. Κυρίες και κύριοι, η UNESCO και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις κίνησαν ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων θεματικών διαδρομών από χώρα σε χώρα ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι ένα καινοτόμο σχέδιο που μας ενώνει, αλλά και ενώνει μεταξύ τους γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς ευρωπαϊκούς ε, τόπους που είναι γραμμένοι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά για να ενθαρρύνει πολιτιστικές επενδύσεις, να αναπτύξει τη δημιουργική οικονομία και να προωθήσει τα ε, προϊόντα μας. Σε όλη την Ευρώπη 34 τέτοιοι ε, το οποίο έχουν ε, εγγραφεί στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα, Δανία, Πολωνία, Κροατία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Αυστρία, Κύπρο και Ουγγαρία. Με το National Geographic ε, θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου για να δίνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να προγραμματίζει το ταξίδι του σε διάφορες γλώσσες. Θα κινητοποιηθούν εκεί όλοι οι παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων. Ε, οι διάφοροι ευρικοί οργανισμοί, οι ξενοδόχοι και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια ευκαιρία αυτή να αναπτύξουμε ένα διαφορετικό όραμα του τουρισμού. Να μην επικεντρωνόμαστε ε, σε κάποιους μεμονωμένους τόπους που έχουν κάποια ε, συγκεκριμένη εποχή ε, μεγάλη προσέλευση, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ διαφαίνεται η δυνατότητα ενός τεράστιου δυναμικού για να αναπτυχθεί η οικονομία, για να ενισχυθεί η επίγνωση και η συνείδηση ε, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ε, του πολιτισμού και για τη διαφύλαξη των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων. Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχε η παράδοση του λεγόμενου Grand Tour, η μεγάλη περιήγηση στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και ήταν τμήμα της εκπαίδευσης κάθε φωτισμένου πολίτη. Και είμαι πεπισμένη ότι ο τουρισμός σήμερα βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο σταυροδρόμι αυτών των φιλοδοξιών που είναι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές. Αυτό το όραμα εγγράφεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εκφράζεται και από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πολιτισμική διπλωματία που κατατέθηκε πέρυσι, η οποία με τη σειρά της βασίζεται σε εργαλεία και μέσα της UNESCO και ιδιαίτερα τη σύμβαση του 2005 για την ε, πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης. Κύριε Πρόεδρε, αυτό επίσης συνδέεται με τη συνεχή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιζητούμε, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα στις οικονομικές προκλήσεις, αλλά και στην κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης. Πράγμα που είναι ακριβώς το μέγα άλλο ατού ε, της πολιτισμικής βιομηχανίας. Είναι στο πλευρό σας η UNESCO, έτσι ώστε αυτή η φιλοδοξία να μεταφραστεί σε κοιτάσματα θέσεων εργασίας δραστηριοτήτων πολιτισμικής δράσης υπέρ της ειρήνης και της ακτινοβολίας των ευρωπαϊκών αξιών. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γενική Διευθύντρια της UNESCO ευχαριστώ για την ομιλία σας και για τις δεσμεύσεις σας για την προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Δίνω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής και ε, τον κύριο Τάση, έχετε το λόγο, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον κύριο Τάση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειών, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι πρέσβεις. Είναι για μένα τιμή όσο και μεγάλη χαρά ευκαιρία που έχω να συμμετέχω σε αυτή την υψηλού επίπεδου διάσκεψη για τον τουρισμό και να εορτάζω μαζί σας την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Προφανώς δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από την Ευρώπη από τον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που επιφυλάσσει το μέλλον στον τομέα αυτό και στις μυριάδες ε, επιχειρηματιών, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και εκατομμύρια ε, εργαζομένων. Η Ευρώπη είναι ο υπαριθμόν έναν παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. 1,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δραστηριοποιούνται και είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά τους στην οικονομία Μάλιστα σε κάποια νησιά μπορεί ο τουρισμός να αποτελεί μέχρι και το 70% του ε, εισοδήματος. Ωστόσο, παραμένουν δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την αστάθεια των τουριστικών ε, ροών, με την ψηφιοποίηση και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδέονται με την συνεργατική οικονομία. Καθώς επίσης και το ε, συνεχές αίτημα βελτίωσης ε, των παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος υπάρχει και η μεγάλη ε, ο μεγάλος ανταγωνισμός από άλλους μη ευρωπαϊκούς ε, προορισμούς. Σήμερα γίνεται λόγος για μαζικό τουρισμό και για σημαντική συγκέντρωση των τουριστών στον ίδιο τόπο. Πράγμα που μπορεί να οδηγήσει δυστυχώς, και το είδαμε συχνά το τελευταίο καιρό, σε εντάσεις μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού και των τουριστών. Για το λόγο αυτό λοιπόν ε, χρειάζεται ένας τουρισμός πιο υπεύθυνος που να σέβεται την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, Αυτό είναι ο σωστό δρόμο να ακολουθήσουμε. Ε, στα πλαίσια αυτά ήδη γνωρίζουμε κάποια καλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η ε, πρωτοβουλία Ευρωπαϊκός Προορισμός ε, Αριστείας. Έχουμε νέους προορισμούς αναδυόμενους ή λίγο γνωστούς, λιγότερο γνωστούς, που σέβονται την αηφορία και τη βιωσιμότητα υπάρχει και ένας ε, κατάλογος βιώσιμος και οικολογικός και όπου υπάρχει ένα eco-label, ένα οικολογικό σήμα που αφορά τα καταλήμματα. Ε, θα πρέπει όμως να ε, συνειδητοποιήσουν την κατάσταση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι ίδιοι ταξιδιώτες, οι τουρίστες, δηλαδή όλοι μας. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι συμπεριφορές μας και οι επιλογές μας για τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και καταναλώνουμε για να ε, σώσουμε την ήπειρό μας, τους κατοίκους και τον πολιτισμό τους. Για να αλλάξουν οι συμπεριφορές, οι δημόσιες αρχές έχουν διάφορων τύπων εργαλεία ε, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση οικονομικά κίνητρα, ε, νομοθεσία και παραδείγματα. Και όλα αυτά τα εργαλεία όμως έχουν τα όρια τους, ε, γιατί δεν επηρεάζουν πάρα πολύ τις συμπεριφορές και την υπεύθυνη κατανάλωση. Ε, πολύ συχνά μπορεί ο καθένας να συνειδητοποιεί κάποια πράγματα εγκεφαλικά, αλλά να μην αλλάζει την καθημερινή του συμπεριφορά. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια πρωτοβουλία ε, που ανάγεται στο 2000 και έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι συχνά δύσκολο να επιβάλλεις με αυταρχικά μέτρα αλλαγές συμπεριφοράς. Είναι πιο εύκολο, έχει αποδειχθεί, αυτό να έρθει από διάφορες πρακτικές και όχι από αυταρχικά μέτρα, όπως υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που ζητούν από τους πελάτες να κάνουν οικονομία στο νερό, να σέβονται το περιβάλλον, να κάνουν οικονομία στην ενέργεια, στο ρεύμα. Και από ό,τι μαθαίνουμε αυτά λειτουργούν και πιάνουν αρκετά καλά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ε, θαρρύνουμε το θεραπευτικό τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, το ε, ιαματικό, γαστρονομικό, ιστορικό και θρησκευτικό. Διάφορα είδη τουρισμού. Αυξάνονται εδώ οι προκλήσεις και πρέπει να είναι αντίστοιχε και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ε, με ε, καλούς επαγγελματίες, με, με μόνιμες θέσεις εργασίας, με βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών. Αυτό ε, θα βοηθούσε να ταξιδεύουν στην Ευρώπη άτομα της τρίτης ηλικίας ή με αναπηρίες περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τους ανθρωπίνους πόρους χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης στρατηγικό έτσι ώστε να έχουμε μια μόνιμη ροή εργαζομένων με προσόντα που ενδιαφέρονται για μόνιμη ε, θέσει εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύονται οι θέσει εργασία στον κλάδο αυτό που αναπτύσσεται πολύ και έχει και μεγάλο δυναμικό απασχολησιμότητας, ιδιαίτερα των νέων. Θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε οι χώρες μας να εξακολουθούν να είναι ο πρώτος ε, τουριστικός προορισμός παγκοσμία. Α κάνουμε την Ευρώπη ένα ε, προορισμό αριστείας που πραγματικά θα δίνει το παράδειγμα. Πρόσφατα η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή απέφθινε ε, μια έκκληση για να έχουμε μια κοινή ε, στρατηγική διαφήμισης για να διαφυλάξουμε την καλή εικόνα της Ευρώπης και του τουριστικού κλάδου. Παραμένει αυτή η έκκληση ενισχύ. Έχει έρθει η ώρα επιτέλους να μας απασχολήσει και μια πραγματική κοινωνική πολιτική ε, για τον τουρισμό. Και γιατί όχι να συσταθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός τουρισμού με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Σήμερα άκουσα νομίζω ομιλίες που βγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, αρχίζουν από τη δική σας κύριε Πρόεδρε. Αν δεν γίνει πρόοδος τουλάχιστον εκεί, τουλάχιστον προβληματιζόμαστε. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών που λέει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Κοινωνική Εταίρη, η Κοινωνία των Πολιτών. Με δύο λόγια οι πολίτες και εκείνο που αποφασίζουν τελικά οι θύνοντες. Ελπίζω τουλάχιστον στον τομέα αυτό να έχουμε μια γνήσια και αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Βέλα, να χαιρετήσω όλους τους βουλευτές που καταφθάνουν από διάφορα κράτη-μέλη Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Χαιρετίζω επίσης τους πολίτες, τους επισκέπτες που βρίσκονται εδώ και που συμμετέχουν σε αυτή την όλομέλεια. Είναι αφιερωμένοι σε εσά κυρίες και κύριοι που είσαστε καθισμένοι εκεί ψηλά στα θεωρία. Σήμερα υπάρχουν βουλευτές, επίτροποι, επιχειρηματίες, εμπειρογνώμονες που συζητούν το μέλλον του τουρισμού. Είναι ο τομέας που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη απασχόληση για τους νέους τα επόμενα έτη. Και από εκεί και το έργο μας σήμερα, όπως κάθε μέρα, είναι αφιερωμένο σε εσά. Και τώρα, ο κύριος Βέλα, που είναι υπεύθυνο για τα θέματα αλληλείας ε, και θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Προέδρε Ταγιάννη. Επίτροπε, αξιότιμα μέλη, υπουργοί, εξοχότητε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους σας. Πάντα είναι χαρά για μένα να έρχομαι εδώ, αλλά σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Είναι η περίσταση που εορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού με τέτοια διακεκριμένη παρουσία εμπειρογνωμόνων και συναδέλφων σε αυτή την εκδήλωση υψηλού επίπεδου. Είναι ένα θέμα τουρισμός που το το γνωρίζω πολύ καλά, είμαι δύο φορές υπουργό τουρισμού και είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω μεγάλη εμπειρία από μέσα, από τον τομέα αυτόν. Και σαν υπουργό τουρισμού συνάντησα για πρώτη φορά τον πρόεδρο τον κύριο Ταγιάννη όταν ήταν επίτροπος υπεύθυνο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και βλέπω ότι ο τουρισμός ε, τον απασχολεί ακόμα Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο αυτού για την πρόσκληση. Το μήνυμά μου εγκατακλείδει ποιο είναι σήμερα. Τα... Μόνο να κερδίσουμε έχουμε τον τουρισμό. Ε, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναπτύξουμε βιομηχανία ε, βιώσιμη και που θα επεκταθούμε και θα, αυξήσουμε τον τομέα ε, βιώσιμα. Εγώ δεν θα τους αποκαλούσα τους υπουργούς μας υπουργού τουρισμού, αλλά υπουργού βιώσιμου τουρισμού, αν εξαρτιόταν από μένα. Θα ακούσουμε πολλούς αριθμούς, στατιστικά στοιχεία, αλλά ένα γεγονός σίγουρα θα ξεχωρίσει. Ότι η Ευρώπη είναι, κινείται προς τον να είναι υπαριθμόν ένας προορισμός τουριστικός, συμβάλλει πολύ στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουρισμός και παρέμεινε αρκετά ανθεκτικός τομέας και πιο σημαντικό το Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος προβλέπει ότι ο τομέας θα, αυξάνεται, ε, θα αυξηθεί τα επόμενα έτη κατά 30%. Όμως το 2030 θα περιμένουμε 800 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Αυτά τα θετικά μηνύματα δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Αντιθέτως, θα πρέπει να σχεδιάσουμε με αποτελεσματικό τρόπο το μέλλον και να ετοιμάσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για τις πολιτικές. Διότι ο τουρισμός έχει τα υπέρ και τα ωφέλη που είναι κυρίως οικονομικά, έχει όμως ε, και κόστος που είναι κυρίως περιβαλλοντικής φύσεως. Άρα θα πρέπει να αποφύγουμε την υπονόμευση των ωφελών που καθιστούν τόσο ελκυστική την Ευρώπη και θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να ρεχιστοποιήσουμε το κόστος. Ένα πρόγραμμα για βραχυπρόθεσμο κέρδος δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ε, μακροπρόθεσμο όραμα, ούτω ώστε να δώσουμε καλύτερη εικόνα της Ευρώπης. Και έτσι δεν μπορεί να είναι ε, δευτερευούση σημασία στο περιβάλλον. Είναι κλειδί για την επιτυχία μας και θα πρέπει η ονομασία της Ευρώπης στον τουριστικό τομέα να ξεχωρίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό λόγω της ποιότητας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουμε η πιο οικολογικά φιλική ε, περιοχή του κόσμου για τον τουρισμό. Απευθύνω έκκληση προς τον τομέα και που τους διαμορφώνονται στην πολιτική. Σας παροτρύνω, παρακαλώ να είσαστε ενεργοί, να δράτε και όχι να αντιδράτε όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ήδη έχουμε καλά παραδείγματα και μοντέλα που δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν σταθερές πρακτικές επιχειρηματικές. Χρειαζόμαστε όμως μία νέα αντίδραση, ούτω ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον και το φυσικό μας κεφάλαιο. Και αυτό πάντα αναλαμβάνεται υπόψη και έτσι να προστατεύουμε και τον τουρισμό. Να θυμόμαστε ότι οι τουρίστες γνωρίζουν και υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα. Οι τουρίστες περιμένουν ε, μια ε, οικολογική εμπειρία και δείχνουμε μελέτες ότι πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών πιστεύουν ότι οι τουριστικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχουν, να ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Όταν παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που ήδη θέλει ο κόσμος. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα το καθήκον μας και έτσι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας έχει ε, πλεονεκτικό όφελος. Ένας μη βιώσιμος τουρισμός δεν είναι ανταγωνιστικός. Θα ακούσουμε πολλά αυτά, από αυτά τα στοιχεία στις διάφορες ομιλίες. Θα αναφέρω ένα-δύο στοιχεία εν συντομία, πολύ σύντομα. Σαν ε, είπε και η Επίτροπος η κυρία Μπενκόφσκα, Έχουμε το πρόγραμμα COSME για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο συγχρηματοδότησε πάνω από 40 ε, υπερεθνικά τουριστικά προγράμματα που οδήγησαν σε αλλαγές στον τομέα. Ο πρόεδρος κ. Στάσης ήδη αναφέρθηκε στο βραβείο για τον Ευρωπαϊκό Προορισμό Αριστείας ε, που υποστηρίζει λιγότερο γνωστούς προορισμούς που έχουν καταβάλει προσπάθειες για βιώσιμη τουριστική διαχείριση και είναι το μεγαλύτερο τουριστικό βιώσιμο δίκτυο στον κόσμο. Και μη λησμονούμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δικτών Τουρισμού που στηρίζει προορισμούς που θέλουν να βελτιώσουν την βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού. Και το όλο χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντο περιέχει και δύο εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Είμαι σίγουρο ότι τα γνωρίζετε. Το οικολογική το σήμα, το οικολογικό σήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθησυχάζει τους καταναλωτές έχουν εγγύηση ότι οι διακοπές τους δεν κοστίζουν στο περιβάλλον και έτσι βελτιώνεται όλη εμπειρία τους. Το αίμα ε, για τη διαχείριση ε, του περιβάλλοντος βοηθά τις επιχειρήσεις να κινηθούν σωστά, να βελτιωθούν όσον αφορά την εξοικονόμηση της ενέργειας, ε, οικονομία των υλικών, εξοικονόμηση ύδατος. Γίνονται οικονομίες και προστατεύεται και το περιβάλλον και έτσι έχουμε και αύξηση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα οικονομική και περιβαλλοντική. Η πρόκληση ποια είναι, όλα αυτά τα εργαλεία να λαμβάνονται υπόψη στι πολιτικέ. Οπότε χρειάζεται περισσότερε επενδύσει και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν τη σωστή υποστήριξη και θα πρέπει να δίδονται και κίνητρα για τι βέλτιστε πρακτικέ που θα έτσι θα διαδοθούν. Είπα ότι η βιώσιμη χρήση του φυσικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει αντανακλαστικό εντό του τουριστικού τομέα. Η φύση, οι άνθρωποι και η οικονομία θα πρέπει να αλληλοενισχύονται. Η βιωσιμότητα δεν είναι ένα ή, ή, εναλλακτική, αλλά είναι συγχώνευση εποφελής και για τις δύο πλευρές. Οπότε, ας είμαστε σαφείς, το Natura 2000 δεν θα πρέπει να αποκλεί τη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη τώρα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση μέσω του σχέδιου δράσης για τη φύση που υιοθετήσαμε πιο πριν αυτό το έτος. Το σχέδιο, στόχοι του σχεδίου είναι, είναι ότι όταν εφαρμόζεται πλήρως η νομοθεσία για τη φύση ε, τότε έχουμε οικονομική απόδοση και ποιοτικές αποδόσεις για την κοινωνία. Ε, ε, το καλύτερο παράδειγμα είναι οι σε τόποι Natura 2000, εκεί που προστατεύεται η φύση. Και έτσι προστατεύονται και η χλωρίδα και η πανίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα για βιώσιμες δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισμός. Και βιώσιμος τουρισμός μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος για την επίτευξη της ενίσχυσης των διαφόρων πτυχών που ανέφερα. Μετά από 25 χρόνια το δίκτυο Natura 2000 ακόμα δεν έχει δρέψει όλους τους καρπούς για να δείξει πώς το κοινωνικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον στην Ευρώπη είναι αλληλένδετα. Μόνο 50% ε, των τόπων Natura ε, τα χειρίζονται σωστά και ε, δεν, δεν έχουμε την πλήρη απόδοση στον αφορά τις επενδύσεις. Ας αρπάξουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Η παράκτιος, η θαλάσσιος τουρισμός είναι ένα άλλο σημαντικό τομέα που δίνει σχεδόν 3 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και εδώ θα πρέπει να πω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το κλειδί. Γι' αυτό προωθούμε το διάλογο και τις συμπράξεις στους τομείς όπως είναι οι κουραζιέρες και συνδέουμε τους, τις προορισμούς τουρισμού μαζί για να προωθούμε περιφέρειες και για να αντιμετωπίσουμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κουραζιεροπλοίων. Τον επόμενο μήνα η διάσκεψη στη Μάτα για τους ωκεανούς επίσης θέλει να οδηγήσει σε νέες δεσμεύσεις για να εξασφαλίσουμε τη προστασία διαφόρων θαλασσιών περιοχών στον κόσμο έτσι θα στείλουμε ένα θετικό μήνυμα και θα δείξουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να ανθίσει το περιβάλλον που είναι κάτι θεμελιώδες για την πρόοδο στον τομέα. Οι προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές μπορούν να είναι άλλο ένα παράδειγμα της διάδρασης που υπάρχει μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και όφελους ε, για τον τουρισμό. Ε, κυρίες και κύριοι, προχόμενος από τη Μάλτα, από την ίσο της Μάλτας, καταλαβαίνω πλήρως τη σημασία που έχει ο τουρισμός. Όχι μόνο σαν οδηγός οικονομικής ευημερίας, Επίσης όμως σαν μια δύναμη για διασύνδεση και ένωση των Ευρωπαίων και των ε, πολιτισμών της Ευρώπης. Για χιλιετίες ο τουρισμός βοήθησε τους λαούς να συνδέονται και να διαδρούν, να προωθούν ιδέες και να διευρύνονται οι ορίζοντες μέσω φυσικών εμπειριών. Αυτό δεν θα σταματήσει και δεν μπορεί παρά να διευρυνθεί και να αυξηθεί με την ψηφιακή επανάσταση και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ένα από τα θέματα που ρηπαίνουν, ένα από τα προβλήματα που ρηπαίνουν και μολύνουν είναι τα θαλάσσια σκουπίδια και τα παράκτια σκουπίδια, κυρίως τα πλαστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το πρόβλημα, προσπαθεί να το καταπολεμήσει μέσω της κυκλικής οικονομίας, την πηγή του, που αναδιαμορφώνει το βιομηχανικό τοπίο και βελτιώνει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εμφανίζεται σαν προοδευτική ε, και αποτελεσματική σαν Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Ήρθε η ώρα για τολμηρές αποφάσεις και όχι για αρχιπρόθεσμα κέρδη, Θέλουμε βιώσιμο μέλλον που μπορεί να διατηρήσει τον τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του τουρισμού ε, στην πρώτη θέση. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι και ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Ταγιάννη για την υποστήριξή σας. Thank you very much, σας ευχαριστούμε πολύ, Επιτροπέ Βέλα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κύριος Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι Επίτροποι, κύριε Πρόεδρε της ΟΚΕ, εξοχότατοι κυρίες και κύριοι. Ο τουριστικός κλάδος είναι άκρο σημαντικός για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, που εκπροσωπεί η Επιτροπή των Περιφερειών. Ο τουρισμός δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα μέσα από διάφορες άλλες βεβαίως ε, παράγει 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αν προσθέσουμε και τις συναφείς υπηρεσίες και μέχρι το 12% των θέσεων απασχόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ένας ακόμα κλάδος ε, δραστηριοτήτων. Στην Ευρώπη πραγματικά είναι ενταγμένο στον τρόπο ζωής μας και αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα προώθησης των δημοκρατικών αξιών και των ελευθεριών, πάνω στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το να ταξιδεύεις λοιπόν στην Ευρώπη είναι να εκμεταλλεύεσαι τη ζώνη Σέγγεν, ε, τα πλεονεκτήματα του ενιαίου νομίσματος και να βλέπεις πώς σφυριλατείται μια ευρωπαϊκή κοινή ταυτότητα που βασίζεται στην εθνική και ακόμα περισσότερο στην τοπική ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό σήμερα θα ήθελα να τονίσω τα θετικά του τουρισμού, θυμίζοντας στη συνέχεια και κάποια άλλα που μας περιμένουν για να ε, έχουμε μόνιμη και βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να γυρίσω λίγο πίσω. Το 1950 είχαμε 25 εκατομμύρια παγκοσμίω. Πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια λοιπόν ταξίδευαν. Δηλαδή 50 φορές περισσότερο από το 1950. Πάνω από 40% των ταξιδιωτών αυτών επέλεξαν ως προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τις χώρες της και άφησαν 340 δισεκατομμύρια ευρώ συνάλλαγμα. Ε, και μόνο αυτό αξίζει να μας χαροποιεί. Τι κάνει λοιπόν την Ευρώπη τόσο ελκυστική και εγωιτευτική. Ε, δεν είναι ένα και μοναδικό το πλεονέκτημα και το ατού της. Είναι ένα σύνολο, ένα μείγμα στοιχείων. Η αρχιτεκτονική μας και η ιστορική μας κληρονομιά. Οι ε, φυσικοί μας πόροι που τους διαφυλάσσουμε και οι δρυμοί. Οι πόλεις μας, ε, τις οποίες έχουν ε, ε, αποθανατήσει τα μεγαλύτερα συγγραφικά και κινηματογραφικά έργα, οι δημιουργίες, οι καλλιτεχνικές, το folklore και να μην λησμονήσουμε φυσικά τη γαστρονομία μας. Και όπως διαπιστώνετε και εσείς θα μπορούσε να είναι πολύ μακρύτερος ακόμα ο κατάλογος αυτός. Και Εκτός από όλους αυτούς τους συναρπαστικούς τόπους και πίσω από αυτούς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους κάνουν να ζουν, να ευημερούν και τους προστατεύουν. Εξ ονόματος λοιπόν της τοπικής και ε, περιφερειακής αυτοδιοίκησης ε, προχωρούν σε έργα ε, με έμπνευση, με εφευρετικότητα και ζητούν και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταπληκτική δημιουργικότητα ε, καλλιτεχνική και άλλη. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα, μου επιτρέπετε. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός δεν είναι ε, πια ε, θεματικός ε, μάλλον δεν εγγράφεται στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων και λυπάμαι γι' αυτό, έχουν βρει το δρόμο και τον τρόπο οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να αντλήσουν χρηματοδότηση από διάφορους διάβλους και ε, απορροφούν σχεδόν όλα τα κονδύλια. Για παράδειγμα, ε, στην Ουαλία χρησιμοποίησαν το Γεωργικό Ταμείο για την ανάπτυξη της Υπέθρου για τεχνολογίες πληροφορίας έτσι ώστε να προσελκύουν ε, τουρίστες στον αγροτουρισμό. Ε, επίσης, η δορυφορική τεχνολογία για να κάνουν διάφορα κυνήγια θησαυρού, περιπέτειες ε, ή να διαχειρίζονται με οικολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους, στον οικολογικό τουρισμό ή webcams για ε, εικονικές επισκέψεις. Ε, πιο νότια τώρα, μια ισπανική ε, περιφέρεια χρηματοδοτήθηκε από τον ορίζοντα 2020 για να δοκιμάσει και να προωθήσει τις καινοτόμες τεχνολογίες για να έχει ένα κλειστό κύκλο ύδατος για τις τουριστικές εγκαταστάσεις των ακτών της Μεσογείου. Τι εννοώ. Έτσι μειώνεται η χρήση του γλυκού νερού ε, στα ξενοδοχεία και στις τουριστικές εγκαταστάσεις ε, και ανατρέχουν περισσότερο στα υπόγεια ύδατα ή στο ε, νερό της βροχής μετά από επεξεργασία. Βλέπετε λοιπόν ότι βγαίνουμε από την πεπατημένη και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι προορισμοί μας, οι τουριστικοί να είναι πιο όμορφοι και να ζει κανείς καλύτερα είτε είναι επισκέπτης είτε είναι Το 2018 που είναι έτος πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να μας παροτρύνει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Τελειώνοντας, θα αναφέρω δύο έργα προτεραιότητας ε, για να μας απασχολήσουν στη συζήτηση στη συνέχεια. Εάν θέλουμε να αναπτύξουμε ε, ένα βιώσιμο τουριστικό κλάδο, αυτό που χρειάζεται είναι ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης και ρύθμιση των διαφόρων ε, πλατφορμών της συνεργατικής οικονομίας. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να επενδύσουμε στα προσόντα και τις δεξιότητε των εργαζομένων. Είναι ο ακρογωνίο λίθος για να τερματιστεί η επισφάλεια που δυστυχώς πολύ συχνά οργιάζει. Αυτό θα έχει ε, ε, άμεση επίπτωση στην ελκυστικότητα και στην ποιότητα των τουριστικών μας προορισμών. Και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να χαρούμε για την ψηφιακή οικονομία, τη συνεργατική και την οικονομία του διαμοιρασμού που επιτρέπει να ταξιδεύουμε με τρόπο διαφορετικό. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά δικαιώματα, ε, η ζωή του τόπου, η πολιτιστική κληρονομιά που άλλωστε είναι και ο πλούτος της υπήρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την ομιλία σας και τη συνεργασία που έχουν τα δύο θεσμικά μας όργανα. Επόμενος ομιλητής είναι επικεφαλής της αποστολής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία πρέσβης Γιάν Τζου Γιάνγκ. Κύριε Πρόεδρε, εξοχότητε, κύριε, εξοχότητες κύριε Ταγιάννη, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προβουλευτές, εκ μέρους της Κινέζικης Αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προσωπικά, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμότατα για τα εγγένεια αυτής της διάσκεψης υψηλού επίπεδου για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια τεράστια δύναμη καλού ε, στον κόσμο, γιατί δίνει, ε, επιτρέπει την ε, οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη γενικώ ενισχύοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις των λαών. Επίσης, ο τουρισμός ήδη αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και μάλιστα στην πανηγυρική διακήρυξη της Ρώμης το περασμένο Μάιο, οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξαν την πολιτική του τουρισμού τομέα στρατηγικής προτεραιότητας για να εφετηθούν οι, προτε... οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και ε, την οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, στην ε, Κίνα έχουμε 10.000 ε, ε, βιβλία και έχουμε, έχουμε ταξιδέψει και 10.000 μίλια για να υλοποιήσουμε συντονισμένη, ανοιχτή και φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη. Και γι' αυτό αναδείξαμε τον τουρισμό στη στρατηγικό πυλώνα και βασική κινητήριο δύναμη του οικονομικού μας μετα, μετασχηματισμού και της οικονομικής αναβάθμισης. Και ως ε, ε κύριε Αγορά, 135 εκατομμύρια Κινέζοι ταξίδεψαν στον κόσμο το 2015 και εξόδεψαν 261 δισεκατομμύρια δολάρια επισκεπτόμενοι διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Και μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι την επόμενη πενταετία οι Κινέζοι τουρίστες θα φτάσουν στα 500 εκατομμύρια, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για κοινή ανάπτυξη και ευημερία. Η αναγνώριση λοιπόν της σπουδαιότητας του τουρισμού ε, και των τουριστικών ανταλλαγών Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύνοδος ε, ε, Κορυφής του 2019 που θα αναδειχθεί και ως ε, χρονιά τουρισμού διεθνώς, θεωρώ ότι θα επικεντρωθεί σε αμοιβαίως επωφελείς συναλλαγές και πολιτιστική συνεργασία και κατανόηση. Έτσι θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό μιας από τις σημαντικότερες σχέσεις που έχουμε στον κόσμο. Και όχι μόνο από τουριστική σκοπιά, αλλά γενικώ ε, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά και πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτή την ε, επιφανή εκδήλωση καλή επιτυχία, καλή τύχη και προσβλέπουμε σε περαιτέρω υποστήριξη και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προώθηση των κοινών μας στόχων της δημιουργίας ε, μιας παλόμενης τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, υποστήριξης της ανάπτυξης και της άνθησης του τουρισμού. Thank you very much, dear Σας ευχαριστούμε κυρία Πρέσβευστα. Επόμενος ομιλητής είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ε, για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό, κυρία Τάμπατα. It's open, Ralph. You want to speak here? It's possible, eh? No. Caro Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Ταγιάννη, ε, Υπουργοί Πρέσβης, εκπρόσωποι των δικήσεων, αγαπητοί ευρωβουλευτές, ενδιαφερόμενοι και αγαπητοί φίλοι και επιφανείς καλεσμένοι. Αγαπημένη μου οικογένεια του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία μου σήμερα σε αυτή την ευχάριστη εκδήλωση και να μας ευχηθώ όλους χρόνια πολλά. Και να σας πω γιατί ε, μιλώ όρθια. Συνήθως οι ευρωβουλευτές όταν εκφωνούν τις ομιλίες τους στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σηκωνόμαστε όρθιοι. Αλλά στέκομαι σήμερα όρθια και όχι, μιλάω όχι καθιστή γιατί είναι πολύ σημαντική ε, ημέρα και θα ήθελα να σταθώ όρθια απέναντί, απέναντί σας όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό τουρισμό και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στο πλευρό μας. Νιώθω εξαιρετικά υπερήφανη που αποτελώ τμήμα αυτής της πρώτης μείζωνος σημασίας εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τουρισμό και θα ήθελα να επενέσω τον πρόεδρο Ταγιάννη, γιατί πραγματικά ε, ασπάστηκε την ιδέα και αποφάσισε να ε, επιτρέψει την διεξαγωγή των συζητήσεων στην Ολομέλεια και επίσης θα είναι και ο οικοδεσπότη της δεξίωσης που θα ακολουθήσει. Χίλια ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την διοργάνωση αυτή και ως συμπρόεδρος της ε, Διακομματική Ομάδας για την Ανάπτυξη του Τουρισμού τα τελευταία χρόνια έδωσα μάχη για τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων στην Ευρώπη. Γι' αυτό και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που έχω την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω μαζί σα για τον τουρισμό, μαζί σα που είστε από τι κορυφαίε πολιτικέ προσωπικότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με του πολύ σημαντικού και επιφανεί ενδιαφερομένου που έχουμε σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα. Το γεγονό ότι έχουμε πολλού εκπροσώπους από τα θεσμικά όργανα τα Υπουργεία Τουρισμού και την τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει πόσο σημαντικό είναι ο τουρισμός σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κοινωνίας. Γι' αυτό και είναι καθήκον μας, ε, εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρόσωποι των πολιτών, να, δια, να τους διαβιβάσουμε, να τους διαμηνήσουμε τη στράτευσή μας υπέρ του τουρισμού. Είχα προετοιμάσει ένα πολύ ωραίο λόγο γιατί είναι η μέρα εορτασμού σήμερα και είχα βάλει στην ομιλία μου όλα τα ωραία που σκέφτομαι για τον τουρισμό, όλο μου το πάθος, το ζήλο και την προσήλωσή μου στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Αποφάσισα όμως τελικά να παρετηθώ της ομιλίας μου και νομίζω ότι σήμερα, αλλά και γενικώ. έχετε ακούσει πολλές ε, ωραίες ομιλίες και εξομολογήσεις ε, έρωτα για τον τουρισμό. Αλλά τα λόγια ε, είναι αρκετά πια. Χρειαζόμαστε πιο απτές ενέργειες, χρειαζόμαστε έργα και θα ήθελα σήμερα να είναι η μέρα που εδώ, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αποφασίσουμε από κοινού να φέρουμε την επανάσταση και να αλλάξουμε τις προτεραιότητες των δημοσίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας τον τουρισμό, που είναι από τις σημαντικές κινητήρες δυνάμεις της οικονομίας μας, να του δώσουμε επιτέλους τη θέση που του αξίζει. Γι' αυτό και αρχίζω την ομιλία μου. Ε, και θα ήθελα να πω ότι είναι αναφυσβήτητο σήμερα ότι ο τουρισμός είναι από τις πιο υποτιμημένους, από τους πιο υποτιμημένους κλάδους στην Ευρώπη, παρά την τεράστια θεκτικότητά του και τη σταθερή του ανάπτυξη, ακόμη και κατά τις πρόσφατες κρίσεις και τους κραδασμούς που βιώσαμε στην Ευρώπη. Παντού στον κόσμο, ο τουρισμός είναι σημαντικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και μάλιστα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών των κοινοφελών. Ε, πάνω απ' όλα όμως συμβάλλει στη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού, της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και παρόλα αυτά δεν έχουμε ακόμη μια στρατηγική, ούτε καν ένα σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για όλες αυτές τις ε, ε, επενδυτικές προτεραιότητες των χωρών και των περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού. Επιπλέον δεν έχουμε καν ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή για να χρησιμοποιηθεί από τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που αντιπροσωπεύουν τον κλάδο. Θα πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν και να αρχίσουμε να βλέπουμε τον τουρισμό ως ξεχωριστό οικονομικό κλάδο Γι' αυτό και θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις υπέρ αυτού. Γι' αυτό και βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα. Ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσουμε ένα άλμα πρόοδου και από το απλώς αναγνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι επωφελής για τις οικονομίες μας, θα πρέπει να τον ε, φέρουμε στο προσκήνιο πανευρωπαϊκά. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεκτιμήσει τον τουρισμό και να ξε... προβλέψει ξεχωριστέ ε, δημοσιονομικέ γραμμέ γι' αυτό στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε στοχευμένε κοινοτικέ δράσει για θέματα αρμοδιοτήτων μα που θα αντικατοπτρίζουν την ανάγκη μιας οριζόντιας προσέγγισης για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Juncker για τον τουρισμό. Ένα επενδυτικό σχέδιο για τον τουρισμό για να γίνει ο κλάδος αυτός βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό να εκπονήσουμε ψήφισμα ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει περισσότερε δράσει και περισσότερε πρωτοβουλίε. Αν θέλουμε να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στου παριθμών ένα τουριστικό προορισμό του κόσμου, Χρειαζόμαστε τουρισμό που θα συμπεριλαμβάνει την τεχνολογία και τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα ε, με επιτυχία, ώστε να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών και να δώσουμε προοπτικές στους νέους μας που σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω της ανεργίας που τους μαστίζει, αλλά να προσφέρουμε και καλές υποδομές, συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα για όλες τις περιφέρειές μας. Τέλος, θα ήθελα να σας υποβάλω μια πρόκληση εδώ. Ας δούμε αυτή την εκδήλωση σήμερα ως την απαρχή της επανάστασης στον τουρισμό. Και να μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός δεν έχει μόνο οικονομική πτυχή. Αφορά τη φιλοδοξία, τις επιθυμίες και την διαφορετικότητα. Όλα αυτά αποτελούν άλλωστε αξίες του ευρωπαϊκού ε, οράματος. Και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ναύρατσης που στήριξε αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ευρωβουλευτές και όλους τους ε, ενδιαφερομένους που κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναδείξει αυτό το έτος ως έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ελπίζω ότι θα το συνδέσουμε αυτό το έτος και το σχετικό ερτασμό με τον τουρισμό. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία, καλή τύχη ε, και αποτελέσματα στον τουρισμό και ελπίζω στο μέλλον ο τουρισμός να γίνει προτεραιότητα των δημοσίων πολιτικών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και σας περιμένω με ανυπομονησία στη δεξίωση υψηλού επίπεδου στην οποία ε, θα σας υποδεχθώ μαζί με τον ε, Πρόεδρο Ταγιάννη σε 7 στο εστιατόριο των Ευρωβουλευτών. And now the Vice Chair of the Committee on Transport and Tourism. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής ε, Τουρισμού ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, ε, εξοχότατη, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι όλοι εσείς που ανήκετε στη μεγάλη οικογένεια του τουρισμού, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απευθύνει χαιρετισμό ο μιλητής και στα Κινέζικα. Πρόεδρε Ταγιάννη, θα ήθελα εκ μέρους ε, αυτής της μεγάλης οικογένειας και εκ μέρους ε, της Επιτροπής Τουρισμού και Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέλαμε όλοι μας να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι επιτέλους ε, έχει βάλει τον τουρισμό πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του. Ε, οι λαμβάνοντες αποφάσεις, οι άμεσα εμπλεκόμενοι από περιφερειακά κοινοβούλια, από το εθνικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε σκεφτεί κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να συλλογιστούμε και να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε το τι ακριβώς έχουμε επιτύχει. Να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση και αν θέλουμε η βιομηχανία τουρισμού στην Ευρώπη να παραμείνει επιτυχής. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο πρέπει πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε ορισμένα ερωτήματα. Δηλαδή, επιθυμούμε την Ευρώπη να την διατηρήσουμε ως τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Ναι, προφανώς επιθυμούμε να ε, περασπιστούμε τα εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης που προσφέρει ο τουρισμός. Ναι, βεβαίως. Μήπως επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες. Προφανώς. Επιθυμούμε ο τουρισμός να οδηγεί στην ανάπτυξη λιγότερων αντιμένων περιοχών της Ευρώπης. Ναι. Θέλουμε ο τουρισμός να εκπροσωπείται καλύτερα στα μεγάλα προγράμματα ανάπτυξης Ευρώπης. Βεβαίως. Επιθυμούμε οι εθνικές κυβερνήσεις να κατανοήσουν την ε, σημασία του τουρισμού και σε άλλους τομείς, βεβαίως. Και επιθυμούμε άραγε οι δημοσιογράφοι πολλοί, των οποίων βρίσκονται σήμερα εδώ, να προσφέρουν μεγαλύτερο χώρο στον τουρισμό. Και σε αυτό η απάντηση είναι κατεφατική. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι και πολλοί από εσά την καταφατικά. Α προχωρήσουμε λοιπόν σε πιο δύσκολε ερωτήσει. Και ρωτώ, ο τουρισμό εκπροσωπείται σωστά στην ε, μερίσια διάταξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Δυστυχώ, όχι. Το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τουρισμό και εδώ η απάντηση είναι όχι. Είναι φυσιολογικό μόνο μια ε, δεκάδα ανθρώπων να ασχολούνται με τον τουρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όταν ο κύριος Γιούνκερ δεν απαντάει σε καμία επιστολή μας που αφορά σε σημαντικά θέματα του τουρισμού. Όχι. Μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηροί όταν μόνο Πολύ λίγα προγράμματα ε, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΦΣΙ και έχουν σχέση με τον τουρισμό. Όχι, στην αλφή, προφανώς και όχι. Δεν είμαι καθόλου ευτυχής με όλα αυτά, αλλά χαίρομαι που συμφωνείτε όλοι με αυτά τα τόσο δύσκολα ερωτήματα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, η οργάνωση συνεδρίων για τον τουρισμό είναι κάτι πολύ καλό και υποφελές για τον κλάδο. Όμως δεν είναι αυτός ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεν ήρθαμε εδώ για να επιταψιλεύσουμε φιλοφρονήσεις και για να συγκεντρώσουμε ωραία στατιστικά στοιχεία τα οποία θα πάμε μετά να μεταφέρουμε στις πατρίδες μας. Πρέπει να γνωρίζετε και ίσως ο πρόεδρος, ο Αντώνιο, το γνωρίζει και είμαι σίγουρο το γνωρίζει καλά, ότι εγώ ως μέλος των σοσιαλιστών δεν στήριξα τον κύριο Ταγιάν, δεν τον ψήφισα για πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικές ε, πολιτικές οικογένειες και έχουμε διαφορετικές απόψεις για πολλά θέματα. Όμως σήμερα ε, με αυτή την εκδήλωση μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Η ομάδα των σοσιαλδημοκρατών, η ε, το η Φιλελεύθερη, η Πράσινη, η Γκουε, όλοι όσοι βρίσκονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφωνούν ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια συμμαχία για να στηρίξουμε τον τουρισμό. Όχι τη γνωστή συμμαχία που κυβερνά, αλλά μια ουσιαστική μεγάλη συμμαχία. Όλοι λοιπόν μπορούν να επαναλαμβάνουν συνεχώς τα επιχειρήματα γιατί ο τουρισμός είναι σημαντικός. Φτάνει όμως με αυτές τις ε, μεγαλοστομίες. Χρειαζόμαστε πράξεις. Ο κύριος Σταγιάννη ως πρώην επίτροπος της Επιτροπής άφησε ένα σημαντικό κληροδότημα για τον τουρισμό ε, οι άμεσα εμπλεκόμενοι τον θυμούνται με νοσταλγία ε, την εμπειρία του για θέματα τουριστικά και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ε, το ιστορικό αλλά και η καθημερινή σχέση με τους εμπλεκόμενους, με τους φορείς του τουρισμού. Ήμουνα πρόεδρος του Ουγγρικού Συμβουλίου για Τουρισμό και εκεί κάναμε ακριβώς το ίδιο. Έμαθα λοιπόν ότι αν οι πολιτικοί είναι πρόθυμοι να ακούν τα αιτήματα του κλάδου, ε, τότε ε, μπορούν να επιτύχουμε πάρα πολλά. Και γι' αυτό το λόγο εγώ αποκοινούμε πολλούς άλλους αδέλφους, άρα όλοι μας ε, από τότε που ήρθαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο συνεργασίας για τον τουρισμό και επιτύχαμε πολλά. Φέραμε κοντά τους ε, πιο άμεσα, τους πιο δυνατούς ε, για να υπογράψουμε ένα μανιφέστο τουρισμού. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για μια σειρά προγραμμάτων που είναι πολύ πιο φιλόδοξα από παλαιότερα. Και κυρίως είμαστε υπερήφανοι για κάποιες δικές μου πρωτοβουλίες, ε, ας πούμε ενδεικτικά, τη συνεργασία με την Κίνα, η οποία προέκυψε καταρχήν ως ένα μεμονωμένο πρόγραμμα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα συνεχίσουμε διότι 2,5 ε, εκατομμύρια θα πάρουμε από το Κοινοβούλιο για τον τουρισμό. Εξίσου σημαντική είναι η πρωτοβουλία επιτόπου ε, για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω του τουρισμού. Ένα από τα προγράμματά μας που αφορά τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις ευθύους τουρισμού, αυτό θα ξεκινήσει ε, την επόμενη χρονιά ε, θα αφορά τους νέους. Και τέλος θέλω να σας πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τη διάσκεψη των Πρόεδρων και βεβαίως τον ίδιο τον Πρόεδρο που δέχτηκαν μια ειδική συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα ε, στα Ηνωμένα Έθνη το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα ε, σημαντικά αποτελέσματα, αλλά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μόνο και αν υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση των τουριστικών προγραμμάτων. Αν ακούσετε προσεκτικά, κυκλοφορούν φήμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2020 θα έχουν ένα ειδικό φυλάκιο για χρηματοδότηση του τουρισμού. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Το λέω εδώ και πολύ καιρό ότι το μόνο εμπόδιο μπροστά μα για να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα στον τουρισμό είναι η ε, ανυπαρξία προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το να διεκδικούμε με κόπο κάποια κονδύλια για προσωρινά προγράμματα. Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καλύπτουν τις πρωτοβολίες του τουρισμού και να βάλουν τον τουρισμό εκεί ακριβώς που το αξίζει. Σας μιλάω ορμόμενος από την εμπειρία μου. Τίποτα δεν είναι ε, γραμμένο σε πέτρα όσον αφορά την πολιτική. Όλα αλλάζουν και είμαι σίγουρος ότι μετά το 2019, τις εκλογές, ε, μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικές αλλαγές και γι' αυτό συμφωνήσαμε να προωθήσουμε αλλαγές οι οποίες θα εκπροσωπούν τα συμφέροντά μας. Πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη μια νέα επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα είναι αρμόδια μόνο για θέματα τουρισμού. Είναι απολύτως απαραίτητο. Και αυτό παράλληλα με την σύσταση μιας νέας θέσης ενός νέου επιτρόπου που θα είναι αρμόδιος μόνο για θέματα τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος οικονομικός κλάδος στην Ευρώπη και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτο ένας κλάδος τέτοιου μεγέθους να μην έχει τη δική του την εκπροσώπηση σε ανώτατο επίπεδο. Ε, ένας από τους μελλοντικού 27 ε, επιτρόπους θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα του τουρισμού. Βεβαίω η Επίτροπο Μπιανκόφσκα και οι συνάδελφοί τη, η Κρίστα Ερή, Τζούλη, η Λόνα, ο Κάρλο, ε, τα τελευταία χρόνια ε, η Άννα και πολλοί άλλοι αυτοί εργάζονται πολύ καλά αλλά δεν αρκεί αυτό ως Αντιπρόεδρος επιτροπή ΤΡΑΝ, αρμόδιος για θέματα τουρισμού και τη Task Force του τουρισμού, εγώ εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο ε, και στις Βρυξέλλες και αλλού, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ως εκ τούτου, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες κατά τα επόμενα έτη που μπορούμε όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε ιστορία με μεγάλες επιτυχίες. Ε, σήμερα νομίζω ότι βάλαμε τον, το θεμελιώδη λίθο. Ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Vice President. Ευχαριστούμε τον ε,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 μαζί σας τη δική μου συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση, ελπίζοντας ότι έτσι θα συμπληρώσω την συνολική εικόνα. Και θα ήθελα να μιλήσω για τη σχέση μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού. Δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν. Τέσσερις στους δέκα τουρίστες διαλέγουν τον τουριστικό τους προορισμό με βάση το πόσο ελκυστικός είναι από πλευράς ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πολιτιστική κληρονομιά είναι βασική βασικό, βασική πηγή για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς απασχολούνται 300.000 άνθρωποι, ενώ 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται εμέσως με την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό και παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της συντήρησης και των σχεδιασμών εκθέσεων. Ο, αν έχουμε έναν κλάδο πολιτιστικής κληρονομιάς που ανθεί, αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους της ε, οικονομίας. Μιλούμε π.χ. για το σχέδιο, για το design, για την κοσμηματοποιία, για τη γαστρονομία, για τις τέχνες, ε, για τις βιοτεχνίες, για τις ε, ε, ε, μικρές μεταποιήσεις και κατασκευές. Όλα αυτά κάνουν μια περιφέρεια σφίζουσα, πολύ πιο ελκυστική για επισκέπτες και τουρίστες. Άλλωστε όλα αυτά έχουν θετικές επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους, στον κλάδο των μεταφορών, τον κλάδο της εστίασης, ε, των ξενοδόχων, των ξεναγών, των μεταφραστών διερμηνέων. Το βασικό νόημα στο να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης ακριβώς έγκυται στο γεγονός ότι θα πρέπει να είναι αυτή διαθέσιμη για να ε, την επισκέπτεται ο κόσμος και να την απολαμβάνει. Η διατήρηση λοιπόν είναι κοινή ευθύνη η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ρόλο πρέπει να διαδραματίσει και το κεντρικό κράτος και η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε, αυτό είναι σε συμφωνία με τις συνθήκες και σε επόμενη και τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Βασικός μου στόχος για το 2018 που θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι να συγκεντρώσει τα φώτα όλων των προβολέων διότι έχει εγγενή αξία στη δημιουργία, στη σφυριλάτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας διότι μας βοηθά στο να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον αλλά διότι συμβάλλει επίσης και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Μας δίνει την ευκαιρία να διαρευνήσουμε τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού τουρισμού. Μπορούμε να διαρευνήσουμε πώς θα δρέψουμε τα οικονομικά ωφέλη του τουρισμού, διασφαλίζοντας συνάμα ότι αυτό θα είναι βιώσιμο αηφόρες. Η Ευρώπη είναι ένας βασικός τουριστικός προσορισμός, διότι έχει μια απαράμιλη, ασύγκριτη πολιτιστική κληρονομιά. 450 τοποθεσίες είναι εγγεγραμμένες στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ε, οι μισές ε, που από τον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και είναι μόνος του, από μόνος του λόγος αυτός να είμαστε περήφανοι για την πολιτιστική μας κληρονομιά στην Ευρώπη, αλλά να νιώθουμε συνάμα και την ευθύνη να την προστατεύσουμε, να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι όλα αυτά τα μνημεία θα είναι αηφόρα, βιώσιμα σε βάθος χρόνου. Με χαρά μου θέλω να πω ότι η UNESCO είναι ένας από τους βασικούς εταίρους μας για το Ευρωπαϊκό Έτο τους πολιτιστικής κληρονομιάς και θα μας βοηθήσει, θα παίξει σημαντικό ρόλο διότι έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, πολιτιστικών ριζών και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εμείς θα ξεκηρύξουμε την έναρξη του έτους αυτού στο Μιλάνο στις 7 Δεκεμβρίου και ελπίζουμε ο πρόεδρος Ταγιάννη να μας τιμήσει με την παρουσία του. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2018 θα απευθυνθούμε σε όλους τους ανθρώπους από όλα τα μετερίζια, κυρίως τη νεολαία, και θα τους ενθαρρύνουμε να ανακαλύψουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και να εμπλακούν, να συμμετάσχουν ιδιαίτερα στην προστασία και στη διατήρησή της. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα μας δώσει την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε, να προωθήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα, το Creating Europe, το Erasmus Plus, το Horizon 2020. Θα στηρίξουμε τη βελτίωση των υποδομών. Θα στηρίξουμε τις τοπικές αρχές για τη διαχείριση όλων αυτών των θησαυρών. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη ψηφιακή σφαίρα διότι η ψηφιοποίηση τη πολιτιστική χρονομιά είναι απαραίτητη για τη μετάδοση αυτή στις επόμενες γενιές, στο να γίνει πιο προσβάσιμη, να απευθυνθεί σε περισσότερα και μεγαλύτερα ακροατήρια, κάτι πολύ σημαντικό για τον τουριστικό τομέα. Έχω συναντηθεί με τους εθνικούς συντονιστές για το θέμα αυτό και τους βασικούς εταίρους από την Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών. Εκπρόσωποι των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αγράφησαν τα βασικά χρηματοδοτικά προγράμματα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνεργασίας. Οι Ευρωπαϊκές ημέρες τουρισμού έχουν συντευθεί με επιτυχία. Εκεί τονίζονται και προωθούνται οι βασικοί σημαντικοί τομείς πολιτικής που θα είναι προτεραιότητα μας. Το 2018 θα είναι και το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Αυτό θα μας δώσει νέες ευκαιρίες. Βασικό κλειδί για την επιτυχία αυτού του προγράμματος είναι να δράξουμε όλες τις ευκαιρίες, να διασφαλίσουμε ότι η σχέση μεταξύ τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς θρέφεται, καλλιεργείται, γίνεται αντικείμενο βιώσιμης αηφόρου διαχείρισης και το 2018 και μετά από αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι όσο σημαντικός και αν είναι ο τουρισμός, ε, το πολύ βλάπτει πάντοτε. Όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ροές ανθρώπων. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ε, υδάτινους πόρους, στη διαχείριση των αποβλήτων, στο σύστημα μεταφορών. Υπερφορτώνονται οι τοπικές κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες και γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ προσεκτικό σχεδιασμό για να μην χάσουμε σε βάθος χρόνου την ανταγωνιστικότητά μας. Να λειτουργήσουμε έξυπνα και να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της εκάστοτε. Γίνεται όμως και θα, είναι, ε, θα υπάρχουν ωφέλη για όλους. Υπάρχουν καλά παραδείγματα που ε, πρέπει κανείς να παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, η πόλη της Μπρίζου στο Βέλγιο. Ε, κάθε φορά γίνεται διαβούλευση με τους πολίτες ε, για, σε κάθε νέα ιδέα, έτσι ώστε να είναι βέβαιες οι τοπικές αρχές ότι κάθε τουριστική δραστηριότητα θα εντάσσεται στην τοπική κοινωνία, στη ζωή της κοινότητας και δεν θα αποτελεί τροχοπέδι στην καθημερινότητα των πολιτών. Και έτσι ένας προορισμός γίνεται πιο ελκυστικός και για επισκέπτες και για πολίτες. Αλλά και στη Φιλανδία έχουμε παραδείγματα όπου ε, οι τοπικές ε, κοινωνίες βρίσκονται στο επίκεντρο της, του, τουριστικού προϊόντος και ε, είναι πάρα πολλοί οι εταίροι που συμμετέχουν στα κοινά προγράμματα και στα κοινά εγχειρήματα. Ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν στο πλαίσιο αυτό του προγράμματος εργασίας για τον πολιτισμό 2015-2018 να ορίσουν εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν πάρα πολλές χώρες, συμμετέχουν και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όπως η Ισλανδία και θα εξετάσουν αυτή τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και αηφορίας και βιωσιμότητας. Και τα ευρήματα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 2018. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι μοναδική κυρίες και κύριοι διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μας βοηθά να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Ε, ε, καλλιεργεί διάφορες δεξιότητες και ε, βοηθάει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη πόλεων, πολιτών και περιφερειών. Δεν έχει σχέση μόνο με το παρελθόν, έχει άμεση σχέση με τη δημιουργία της Ευρώπης του αύριο. Και γι' αυτό διαλέξαμε το εξή σλόγγαν η κληρονομιά μας. Εκεί όπου το παρελθόν συναντάται με το μέλλον. Αυτή θα είναι, αυτό θα είναι το μότο, το βασικό σλόγγαν για το 2018, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά την επόμενη χρονιά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, σας προσφέρει στήριξη στο πολύ σημαντικό σας έργο. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Θα ήθελα τώρα να σας ε, δώσω δύο-τρεις ενημερωτικές πληροφορίες. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού θα προεδρεύσει στην επόμενη στρογγυλή τράπεζα πώς θα προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, θα βελτιώσουμε τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό κλίμα. Σας παρακαλώ λοιπόν τώρα να σηκωθείτε. Θα έχουμε μια οικογενειακή φωτογραφία για να ε, παραμείνει, να παθανατιστεί αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, ε, τα στελέχη, τα μέλη του δικού μου του γραφείου που κατέστησαν δυνατή αυτή τη σημερινή ημερίδα που ήταν πάρα πολύ σημαντική για να δώσουμε όθηση στον τουρισμό στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας.